Bien. Buenas tardes. Vamos a, dar comienzo. Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε αυτή την ε, συνεδρίαση εργασίας για την αγορά ε, ενέργειας, τη ρύθμιση, τα τιμολόγια ενέργειας. Πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία να συζητήσουμε μεταξύ ευρωκοινοβουλευτικών και εθνικών κοινοβουλευτικών αυτό το ζήτημα. Τα αγγλικά δεν λειτουργούν, λέει η Πρόεδρος. Repeat no? Sí. Λειτουργούν τα αγγλικά τώρα, θαυμάσια. Έλεγα ότι είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα It's Έλεγα ότι είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε για την ενιαία αγορά ενέργειας, τη ρύθμιση και τις, ε, τα τιμολόγια ενέργειας. Γι' αυτό μαζί με την Πρόεδρο και με τον κύριο Λαβίγια, ο οποίος είναι από το Ισπανικό Κοινοβούλιο, θα συζητήσουμε επίσης εδώ και ο κύριος Ρότε Στράους, ο οποίος θα λάβει και αυτό το λόγο και στη συνέχεια θα υπάρχει δυνατότητα να θέσετε ερωτήματα, να ξεκινήσουμε μια συζήτηση και εάν θέλετε να λάβετε το λόγο παρακαλούμε να αναφέρετε και το όνομά σας για να μπορούμε να γνωρίζουμε και ποιοι είσαστε. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην σύντροφο Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Σύντροφε, αν μπορώ να το πω έτσι. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε όλοι σας. Στην συνεδρίαση αυτή για την ενιαία αγορά, τον ανταγωνισμό και την ενέργεια. Μαζί με την Μαρισκα από την ε, γερουσία τη Ισπανίας έχουμε έρθει και περισσότερο τον κύριο Μαρτίνες που είναι συγητής για την ομάδα μα Τα θέματα λοιπόν που θα μας απασχολήσουν εδώ έχουν ε, αποτελέσει κέρια θέματα στην ευρωπαϊκή κοινότητα ήδη από την ΕΚΑΧ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι αρμοδιότητες όμως για μια συνολική πολιτική για την ενέργεια απέδειξαν στη δεκαετία του 70 αποτυχημένες. Μπορέσαμε αργότερα όμω και 30 χρόνια αργότερα στη συνθήκη τη Λισαβόνα να έχουμε ένα άρθρο για κοινή πολιτική, για συναπόφαση, που πάλι δεν είναι αρχική. Έχουμε τρει ομάδε εργασία με μια καλή δομή, κατάλαβα μια καλή δομή των προκλήσεων που αντιμετωπίσουμε, στον τομέα της ενέργειας. Η ομάδα μα, η ομάδα εργασία δηλαδή, θα επικεντρωθεί στο τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις πατρίδες μας, για να ενισχύσουμε την ε, ασφάλεια στην προμήθεια ενέργειας, να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να προσφέρουμε όσο περισσότερα μπορούμε, όσο τις υπηρεσίες μπορούμε και καλύτερες για τους καταναλωτές με μια εσωτερική αγορά της ενέργειας. Έχουμε αρκετά νομοθετήματα λοιπόν που έχουμε υιοθετήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκ των οποίων το πιο πρόσφατο ήταν το τρίτο ενεργειακό πακέτο μέτρων πέρσι υιοθετήθηκε. Ωστόσο παρουσιάζονται προβλήματα ως προς την υλοποίηση και τις, τις προηγούμενες νομοθετικών μέτρων. Αφενός. Αφετέρου, η πολιτική ανταγωνισμού μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Πλην όμω με πολύ υψηλή συγκέντρωση αγορέ στην Ευρώπη και περιορισμένη ανάπτυξη δραστηριοτήτων πέραν των συνόρων από του παρόχου, ε, οι οποίοι εξαρτώνται από τις ε, εθνικές τους κυβερνήσεις, δεν υπάρχει επαρκής πρόοδος. Η φορολογία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα θετικό κίνητρο που και πάλι όμως ανήκει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Με αυτά τα τρία στοιχεία ως γνώμονα μπορούμε να ξεκινήσουμε την διερεύνηση του πώς μπορούμε σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας έτσι ώστε να αναπτύξουμε μια πραγματική εσωτερική αγορά αποτελεσματική που να προσφέρει πραγματικές επιλογές και καλές τιμές για τον καταναλωτή. Περιμένουμε από εσά τις συνεισφορές σας, οποίες θα λάβουμε με πολύ προσοχή υπόψη, καθώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ στόμα θα αρχίσει να επεξεργάζεται μια έκθεση για ένα πρόγραμμα δράσεω 2011-2020, πολιτέ πρόγραμμα, και επίσης προσμένουμε να δούμε και πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον της των Ευρωπαϊκών Υποδομών Ενέργειας. Δίνω το λόγο λοιπόν στον εισηγητή εκ μέρου ομάδα μας, τον κύριο Λαβίρνα Μαρτίνε, για να μα κάνει την εισήγηση στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι μας φαίνονται πολύ ενδιαφέρουσε οι συζητήσεις που έχουμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε αυτές τις ημέρες με συμμετοχή όλων των κρατών. Έχουμε την προσπάθεια να, ανα, να ξεκινήσουμε να οργανώσουμε μια εσωτερική αγορά της ενέργειας, μια ενέργεια πιο αηφόρο με τιμές πιο καλές, με πολύ καλές διασύνδεσεις, γιατί χωρίς διασύνδεση ικανοποιητική δεν μπορούμε να έχουμε το εσωτερική αγορά ούτε ανταγωνιστικότητα στην ενέργεια. Και άρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στον 21ο αιώνα. Μπορεί λοιπόν η Ευρώπη, χρησιμοποιώντα ε, πιο αποτελεσματικά του ενεργειακού πόρου, να αποτελέσει τον πρωτοπόρο στην υπόθεση αυτή. Η Ευρώπη έχει ήδη αναπτύξει μεγάλη πρωτοβουλία στην ε, πολιτική αυτή και μπορούν, μπορεί να αναπτύξει το γενικότερο πλαίσιο για την ενεργειακή πολιτική ήδη από την Κοπενχάγη φαίνεται, από τη διάσκεψη του Κοπενχάγης φαίνεται ότι θα πρέπει εμείς να ορίσουμε ποια είναι, ποιοι είναι οι στόχοι για την ενεργειακή πρόοδο για να μην χάσουμε την πρωτοπορία. Πρωτοπορία τι σημαίνει, σημαίνει και κοινοτομία, σημαίνει και δημιουργία νέων συνεργασία και θα πρέπει η Ευρώπη να δείξει πώ εξασφαλίζεται προμήθεια σε ενέργεια αποτελεσματικά και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Οι ανανεώσιμε πηγέ ξεκίνησαν, μάλλον παραγνωρίστηκαν στη δεκαετία του 1980 και αυτό στρατηγικό σφάλμα. Αυτό μπορούμε λοιπόν να το διορθώσουμε μόνο εφόσον η επιχειρήση αλλά και ο ιδιώτης, ο καταναλωτής μπορεί να έχει υπαρκούς ε, ποιότητα ενέργεια σε καλές τιμές. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη να υπάρξει ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό μπορεί να βασιστεί στη δημιουργία δικτύων ενέργειας για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους της ενεργειακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εξοικονόμηση ενέργειας, η επίτευξη των στόχων ενέργειας, η αποδοτικότητα, η μείωση της εκπομπής διοξιδίου του άνθρακος, η βιωσιμότητα λοιπόν και η ασφάλεια για την τροφοδοσία, όλα αυτά θα δημιουργήσουν ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι θετικό για τις εξωτερικές ε, σχέσεις επίσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται ένα μεγαλύτερο επίπεδο διασύνδεσης των δικτύων ενέργειας και μια διαφοροποίηση των παρόχων ενέργειας. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα μιας Ευρωπαϊκή Υπήρου που δεν έχει μεγάλες πηγές ενέργειας δικές της. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διατρέξουμε για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο καθαρής ενέργειας, σε επαρκές επίπεδο, αλλά η Ευρώπη πρέπει να παίξει ένα πρωτοπόρο ρόλο στο να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Οι πρωτοβουλίες για τη διασύνδεση δεν έχουν ακόμα κακοφορήσει πλήρω. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την σωστή χρηματοδότηση των υποδομών, δεδομένου ότι η αγορά από μόνη τη δεν μπόρεσε να επιτύχει αυτό το στόχο για το σύνολο τη Ευρώπη η τωρινή οικονομική κρίση μας καταδεικνύει ποια είναι τα αποτελέσματα της έλλειψης ρύθμισης για τα θέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σαφώς έχει την υποχρέωση να παρέμβει για να υπερπηδηθούν όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία μας εμποδίζουν να φτάσουμε το στόχο μιας κοινή αγοράς σε ό,τι αφορά την παροχή ενέργειας. Χωρίς συνδεδεμένα δίκτυα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι της αλληλεγγύης, της ασφάλειας εφοδιασμού και της ανταγωνιτικότητας. επίσης η επίτευξη των στόχων σε ανανεώσιμες ενέργειες και εναντίον της κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει λοιπόν να περάσουμε από τη συζήτηση στην πράξη, από τη θεωρία στην δράση. Η Ευρώπη δεν μπορεί να περιμένει σε μια στιγμή που αλλάζουν πολλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό εμείς θα πρέπει να στοχεύσουμε στην καλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της χρήσης ενέργειας, ε, κάτι που θα μας δώσει τη δυνατότητα να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Με μια αγορά ενέργειας που βασίζεται στη διασυνδέση μπορούμε να αναπτύξουμε και τις ανανεώσιμες ενέργειες. Η ενέργεια δεν έχει σύνορα και πρέπει να υποστηρίζει όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Με ένα διασυνδεδεμένο πλαίσιο ενέργεια, όλα αυτά θα γίνουν πραγματικότητα. Πρέπει επίση να λάβουμε υπόψη το γεγονό ότι ο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών έχει τονίσει ότι υπάρχει 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπων στον κόσμο που δεν έχουν ακόμα ηλεκτρική ενέργεια. Αν η Ευρώπη μπορεί να είναι πρωτοπόρο τη καινοτομία για τη βιώσιμη ενέργεια, μπορεί να είναι το σημείο αναφορά για τι χώρε αυτέ για να μπορέσουν να επιλύσουν τα προβλήματα ενέργειά του. Και θα ανοίξουν έτσι αγορέ. Μία αγορά ενέργειας η οποία καταναλώνει λιγότερο και παράγει περισσότερο δεν θα επιβαρύνει τις νέες γενιές και θα είναι πιο ανταγωνιστική και επομένως θα είναι σε θέση να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Υπάρχουν λοιπόν ισχυροί λόγοι οι οποίοι συνηγορούν υπέρ μιας κοινή αγορά ενέργεια, αλλά πρέπει να περάσουμε και στην πράξη η Ευρώπη του 27 θα πρέπει να συνεχίσει να προχωρεί προς μια κοινή δράση γιατί βρισκόμαστε ενώπιον μιας παγκόσμιας κατάστασης όπου η κρίση στα χρηματοοικονομικά μας κάνει υποχρεωμένους να δράσουμε στον τομέα αυτό. Πρέπει να στοχεύσουμε στις ανανεώσιμες ενέργειες που είναι το μέλλον της Ευρώπης και όλη του κόσμου και αυτό θα οδηγήσει στην ανθρώπινη ευμάρεια και στην προστασία του περιβάλλοντος. Θα είναι η καλύτερη κληρονομιά που μπορούμε να δώσουμε στις επερχόμενες γενιές. Αυτά. Gracias, Feliz. Ε, ευχαριστώ. Ο κύριος Ρόλφ Στράουχ θα λάβει το λόγο τώρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσω τα μέτρα στήριξης τα οποία κυκλοφόρησε η τράπεζα σήμερα μάλιστα επίσημα σε αυτές τις εκθέσεις ε, σε αυτές τις εκθέσεις λοιπόν για τις αγορές ε, ενέργειας και για την οικονομία της αγοράς εξετάζουμε το θέμα φυσικά από την πλευρά της αγοράς, από την πλευρά την νομισματική, από την πλευρά την πιστοτική Παρ' όλα αυτά διαμορφώνουμε μια ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο οι αγορές ενέργειας επηρεάζουν τον πολίτη και επηρεάζουν και την δυνατότητα του πολίτη να καλύπτει τις ανάγκες του σε ενέργεια και οικονομικά βέβαια. Εξετάζουμε ορισμένα στρατηγικά χαρακτηριστικά των αγορών αυτών τα τελευταία χρόνια. Εξετάζουμε την ε, σε επιπτώσεις τις οποίες έχουν οι τιμές των καυσίμων στην πραγματική οικονομία, πώς οι τιμές των καυσίμων επηρεάζουν την πραγματική οικονομία και προσπαθούμε να δούμε πόσο επηρεάζουν πολύ πιο συγκεκριμένα τον πληθωρισμό, σαν παράδειγμα, τις πληθωριστικές τάσεις, οι τιμές της ενέργειας. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε εδώ ένα πλαίσιο αναφοράς σχετικά με τις, ε, το πόσο επηρεάζουν οι τιμές της ενέργειας στον πληθωρισμό. Βλέπουμε πως έχει λειτουργήσει στο παρελθόν, βλέπουμε το πρώτο επίπεδο επιπτώσεων και το δεύτερο επίπεδο επιπτώσεων. Το πρώτο επίπεδο επιπτώσεων είναι άμεσα το ύψος της τιμής το ύψος της τιμής επηρεάζει τον χρήστη και τις τιμές τις οποίες έχει στη διάθεσή του ο χρήστης. Και ταυτόχρονα η ανταπόκριση του χρήστη επηρεάζει το επίπεδο της κατανάλωσης. Το δεύτερο επίπεδο, το δεύτερο επίπεδο επιπτώσεων είναι ο ρόλος τον οποίο παίζουν οι τιμές της ενέργειας στην περίπτωση όπου υπάρχουν έντονες πληθωριστικές τάσεις. Καταρχάς, η, ποιος είναι ο ρόλος της τιμής των καυσίμων. Βλέπετε εδώ στον πρώτο πίνακα τη συνεισφορά των διαφορετικών συνιστοσών των τιμών των υγρών καυσίμων και τις εξελίξεις των τιμών τα τελευταία χρόνια. Εδώ βλέπουμε ότι η βασική πηγή των αυξήσεων των υγρών καυσίμων για τον καταναλωτή τα τελευταία χρόνια είναι η τιμή του πετρελαίου, του αργού που έφυγε από τα 10 σέντ και έφτασε το 140 και το 2008. Αν δει κανείς τα περιθώρια κέρδους που έχουν τα δηληστήρια ή οι διανομής της, του πετρελαίου και των υγρών καυσίμων, εκεί δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα και τα ποσοστά αυτά παραμένουν περίπου σταθερά. Ο δεύτερος παράγων και πιο σημαντικός καθοριστικός παράγων της τιμής φυσικά. Βλέπετε ότι οι φόροι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και επηρεάζουν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο παράγοντα την τιμή και οι φόροι είναι και αυτοί οι οποίοι εξηγούν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τις διαφορές της ε, τιμής των υγρών καυσίμων. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς από την τιμή του δηληστηρίου φτάνει κανείς στην τιμή του καταναλωτή. Μία αύξηση 10 σέντ, 10 λεπτών στην περιοχή του ευρώ προσπαθούμε να υπολογίσουμε πόσο φτάνει στον τελικό καταναλωτή. Το πέρασμα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Το 50% της αύξησης της τιμής χρειάζεται δύο εβδομάδες για να περάσει στον καταναλωτή και το 90% χρειάζεται τρεις με έξι εβδομάδες από τη στιγμή που αυξηθεί δηλαδή η τιμή του πετρελαίου, του καυσίμου αυτή τη στιγμή παράγεται από το δηληστήριο. Και εδώ η ανταπόκριση είναι πολύ πιο γρήγορη όταν υπάρχουν αυξήσεις της τιμής από ότι όταν υπάρχουν μειώσεις της τιμής. Πέρα από το υγρά καύσιμα, ας δούμε τώρα ένα δεύτερο σημαντικό συστατικό των τιμών ενέργειας όπως αυτό εκφράζεται μέσα από τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο 2,3 και 1,8 του συνόλου. Όπως βλέπετε εδώ στο πρώτο διάγραμμα, το επίπεδο της τιμής του ηλεκτρισμού στην περιοχή ευρώ, η διάσπαση της τιμής δηλαδή οι ανώτερες και οι κατώτερες τιμές που βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ μεγαλύτεροι στον ηλεκτρισμό από ό,τι στο φυσικό αέριο. Στο φυσικό αέριο οι διαφοροποιήσεις στις τιμές είναι πολύ μικρότερες από ό,τι στον ηλεκτρισμό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό βέβαια σχετικά με τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο Προσπαθούμε να εξηγήσουμε το τι διαμορφώνει τις ε, διαφορές αυτές. Προφανώς οι φόροι Προφανώς όμως και η ανταγωνιστικότητα και τα επίπεδα αποτελεσματικότητας του δικτύου διανομής. Βέβαια οι φόροι παίζουν ρόλο εδώ αλλά όχι τόσο σημαντικό όσο στα υγρά καύσιμα γιατί οι φόροι στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ μικρότερη ποσοστιαία σε σχέση με τα υγρά καύσιμα. Το επίπεδο λοιπόν του επιπλέον κόστους από όλα τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του όπως διαμορφώνεται είναι μικρότερο από το αντίστοιχο επίπεδο των υγρών καυσίμων. Τώρα, οι αγορές ενέργειας και ο ανταγωνισμός. Έχουμε ήδη συζητήσει το θέμα στο παρελθόν. Υπάρχουν δυσκολίες ως προς το διορισμό της ανταγωνιστικότητας. Υπάρχουν de jure και de facto διαφορές. Ο ανταγωνισμός της αγορής ενέργειας είναι δύσκολα υπολογίσιμος. Υπάρχουν επίσης και κάποια τμήματα της αλυσίδας διανομής τα οποία ουσιαστικά συνιστούν αυτό το οποίο οικονομικά ονομάζουμε ουδέτερα μονοπόλια. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχει υπάρξει αρκετά σημαντική ε, πρόοδος σε σχέση με τη ρύθμιση των αγορών. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα περιθώρια ανταγωνισμού και το λεγόμενο unbundling της ιδιοκτησίας των δικτύων, δηλαδή μια διάσπαση της ε, ιδιοκτησίας των δικτύων. Συνήθως ε, υπάρχουν τρεις εταιρείες, δύο με τρεις, οι οποίες κυριαρχούν στην αγορά αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το ε, αλλάξουμε μέσω της λεγόμενης λοιπόν αποδεσμοποίησης ε, ή του unbundling. Αυτό ισχύει φυσικά για τα υγρά καύσιμα κυρίως και λιγότερο ισχύει για το φυσικό αέριο και για τον ηλεκτρισμό. Βλέπουμε τα ποσοστά των δύο ή τριών μεγαλύτερων επιχειρήσεων που φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις, στο φυσικό αέριο σαν παράδειγμα, σε πάνω από το 70% του συνόλου του διακινούμενου προϊόντος. Η, φιλελεύθερη, η φιλελευθεροποίηση των αγορών βοηθάει ε, την διαμόρφωση των τιμών έχει βοηθήσει η απελευθέρωση της αγοράς στο να κατέβουν οι τιμές για τον καταναλωτή, ιδιαίτερα στον τομέα του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου. Για την περιοχή ευρώ που είναι με, τις, με το μπλε χρώμα αντίθετα από τον υπόλοιπο κόσμο, η έλλειψη φιλελευθεροποίησης έχει αυξήσει κατά 10% τις τιμές. Συνεπώς η απελευθέρωση των αγορών συστηματικά λειτουργεί υπέρ των συμφερόντων του καταναλωτή. Ένα από τα επιπλέον σημεία το οποίο έχει ξεκαθαρίσει σε σχέση με το παρελθόν στον τομέα της ενέργειας, του ηλεκτρισμού, του φυσικού αερίου είναι το πώς περνούν οι τιμές από την παραγωγή στον καταναλωτή αν συγκρίνει κανείς την κατάσταση που υπάρχει ε, για το πέρασμα από τα υγρά καύσιμα στο φυσικό αέριο, η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη και υπάρχει μια καθυστέρηση 6 με 8 μήνες περίπου. Φαίνεται λοιπόν ότι οι αγορές του φυσικού αερίου ανταποκρίνονται με πολύ πιο αργό ρυθμό. Αν κοιτάξει κανείς τον ηλεκτρισμό, υπάρχει μια σαφέστατη διαφορά ανάμεσα στη χονδρική αγορά και την λιανική αγορά σε αυτό το οποίο τελικά καταλήγει στον καταναλωτή δηλαδή. Από την αριστερή πλευρά βλέπετε τις τιμές του πετρελαίου. και την χονδρική τιμή ηλεκτρισμού. Βλέπετε ότι υπάρχει μία διασύνδεση ανάμεσα στα δύο, το ίδιο ισχύει και για το φυσικό αέριο. Στο δεξί διάγραμμα βλέπετε την τιμή του πετρελαίου και την τιμή καταναλωτή ε, ηλεκτρικού ρεύματος στον καταναλωτή. Βλέπετε ότι η τιμή στον καταναλωτή είναι σαφέστατα πολύ πιο σταθερή και δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από τη διακύμανση της τιμής του πετρελαίου. Λόγω ακριβώς του ρόλου που έχουν οι ανταλλαγές αυτές και τα περάσματα από τη μία ενέργεια στην άλλη, έχουν υπάρξει κάποιες διαφορές και στην τιμολόγηση στην συμπεριφορά μάλλον που οδηγεί στις τιμολογήσεις για τα καύσιμα και οι τιμές για τον καταναλωτή πρόσφατα φαίνεται ότι αλλάζουν πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Μέχρι τώρα συζητήσαμε για τις άμεσες ε, επιπτώσεις. Θα θέλαμε να αναφερθούμε λίγο περισσότερο τώρα στις δευτερεύουσες επιπτώσεις. Ο πίνακας εδώ δείχνει ότι οι επιπτώσεις των τιμών του πετρελαίου στον πληθωρισμό διαφοροποιείται από το ύψος της τιμής βέβαια και αυτό είναι κατανοητό εύκολα. Υψηλέ τιμές φυσικά πετρελαίου οδηγούν σε ένα μεγαλύτερο τμήμα της δαπάνης ε, για, ε, του χρήστη για ε, ενέργεια. Συνεπώς η επίπτωση στον πληθωρισμό είναι μεγαλύτερη. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι δευτερεύουσες επιπτώσεις επηρεάζουν κατά 50 περίπου τις 100 τον τρόπο με τον οποίο η ενέργεια επηρεάζει τον πληθωρισμό. περνάει μέσα από αυξήσεις τιμών γενικότερα στην αγορά, από τον καθερισμό του ύψους των τιμών αυτών σε διάφορες δραστηριότητες και προϊόντα. Και αν προσπαθήσουμε να αποσυνδέσουμε εμείς τις επιπτώσεις των μισθών, των αμοιβών, βλέπουμε ότι η αντίδραση των αμοιβών σε σχέση με τις διακυμάνσεις της τιμής της ενέργειας επηρεάζουν και αυτές με ε, αρκετά σημαντικό τρόπο τον πληθωρισμό, τις πληθωριστικές τάσεις. Αν το δει κανείς ε, νομισματικά και μακροοικονομικά, διαπιστώνει ότι η πολιτική που παρακολουθεί αν θέλετε τις εξελίξεις αυτές δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολύ τίποτα σε σχέση τουλάχιστον με τις πρωτογενείς επιπτώσεις. Αλλά παρόλα αυτά σε σχέση με τις δυνατότητες σταθεροποίησης των τιμών και των προσδοκιών για τη σταθεροποίηση των τιμών, να μην επηρεάζονται δηλαδή άμεσα και γρήγορα από τις διακυμάνσεις των αγορών, και εννοώ των αγορών ενέργεια. Αυτή είναι η προσπάθεια την οποία κάνει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την τελευταία δεκαετία. Η ευθύνη αυτή φυσικά δεν ανήκει μόνο σε αυτούς στις τράπεζες, στην κεντρική τράπεζα ή στις κεντρικές τράπεζες, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι καθορίζουν τα ύψη των αμοιβών και την ικανότητα γενικά της περιοχής του ευρώ και των οικονομιών της περιοχής του ευρώ να αντιμετωπίζουν και να απορροφούν με πιο ε, ομαλό τρόπο τις αυξήσεις της τιμής της ενέργειας διαμορφώνοντας κάποιες διαρθρωτικές πολιτικές κατάλληλες για τις ανάγκες της κατανάλωσης η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα της οικονομίας της ζώνης του ευρώ είναι απαραίτητες για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις των διακυμάνσεων των τιμών της ενέργειας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρότ. Μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε το γύρο ερωτήσεων και παρατηρήσεων. Ο κύριος έχει ζητήσει το λόγο ήδη από την Ιρλανδία. Ναι, ναι, ζητήσατε το λόγο, πράγματι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι μέλος του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου και πρώην βουλευτής εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ορισμένα ερωτήματα και κάποια σχόλια. Καταρχήν για τα θέματα της διασύνδεσης μεταξύ των χωρών. Αυτό είναι φυσικά πάρα πολύ σημαντικό για μας γιατί είμαστε νησί και θα ήθελα να έχω την άποψή σας για το πώς θα πρέπει να χρηματοδοτούνται οι διασυνδέσεις, πώς θα πρέπει να την χάνουν διαχείριση και πώς θα τιμολογείται το κόστος της διασύνδεσης για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια κοινή πολιτική τιμολόγηση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διασύνδεση της ισχύω. Επίσης, νομίζω ότι οι παρουσιάσει μέχρι στιγμή δεν έχουν αναφερθεί καθόλου στα βιοκαύσιμα. Εγώ πιστεύω ότι τα βιοκαύσιμα θα διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο, τουλάχιστον για τη συμπαραγωγή θερμότητος και ενέργεια και επίση στον τομέα μεταφορών τα επόμενα χρόνια. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει και η διαφορετική μεταχείριση των βιοκαυσίμων στι διάφορες χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει κοινή αγορά για τα θέματα αυτά. Η αγορά εθανόλη, παραδείγματο χάρη, σε ορισμένε χώρε καλύπτεται από χαμηλού δασμού. υψηλή δασμή μάλλον για να βοηθηθεί χαμηλότερη δασμή για να ευνοηθεί τοπική βιομηχανία και άλλες έχουν πιο υψηλούς δασμούς. Αν δείτε την Αγγλία και τη Σουηδία έναντι χάρη της Ισπανίας και της Πορτογαλίας βλέπετε ότι υπάρχει μια διαφορά έμφαση σε σχέση με την ε, εσωτερική παραγωγή βιοκαυσίμων ή την εισαγωγή τους. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν υπάρχουν οι χώρες οι οποίες εισάγουν φτηνή εθανόλη για να την ξανά εξαγάγουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο οδηγεί σε <clears throat> αθέμητο ανταγωνισμό στις χώρες που προσπαθούν να κρατήσουν υψηλές τιμές. Επομένως, το θέμα της παραγωγής εθανόλης και βιοδίζελ έχει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι τα σχόλιά σας σχετικά. Επίσης, σε ό,τι αφορά τον διαχωρισμό της ιδιοκτησίας του δικτύου από τη λειτουργία του δικτύου, και από δράσεις επισκευών και αρρωγής. Σε πολλές χώρες <clears throat> έχουμε πολύ σημαντικά κρατικά μονοπόλια, κρατικές εταιρείες που ακόμα είναι κύριοι της ε, ικανότητας παραγωγής και των εγκαταστάσεων. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε την οδό της αποδεσμοποίησης για να υπάρχουν ανεξάρτητα συστήματα <clears throat> τα οποία δεν θα ελέγχονται από αυτούς οι οποίοι παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια. Τέλος, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι εγώ ανησύχησα διότι στην προηγούμενη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δόθηκε μεγάλη έμφαση στο να υπάρξει μια νέα ενεργειακή συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να δαπανίσουμε πολύ χρόνο και πολύ προσπάθεια και πολύ πολιτικό κεφάλαιο προσπαθώντα να καταλήξουμε σε μια νέα συνθήκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενέργεια. Αλλά αυτή η προσπάθεια θα ήταν πιο επωφελή στο να εξασφαλίσει ότι θα γίνουν κάποιε πρακτικέ ενέργειε και θα εδρεωθεί η συνεργασία μεταξύ των χωρών μα βάσει του τωρινού νομοθετικού πλαισίου, δηλαδή βάσει τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Από την οπτική γωνία τη δική μου χώρα και τη γείτονο, θα ήταν πολύ δύσκολο να περάσει οποιαδήποτε νέα συνθήκη μέσα στα επόμενα χρόνια. Παρά το γεγονός ότι μια νέα συνθήκη που θα αφορά την ενέργεια στην Ευρώπη θα ήταν επιθυμητή, από πολιτική άποψη θα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Εγώ θα προτιμούσα να λειτουργήσουμε σε πρακτικό επίπεδο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Ευχαριστώ. Προτού δώσω το λόγο στους συναδέλφους μου στο πάνελ, θα ήθελα να πω σε σχέση με τη διασύνδεση ως μέλος του Ισπανικού Κοινοβουλίου και μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας εκεί, πρέπει να πω ότι στη δική μου χώρα έχουμε μόνο 2,5% της ηλεκτρικής ενέργειας που είναι διασυνδεδεμένη με την Γαλλία, πολύ λιγότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει και προβλήματα ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης της οικονομίας μας λόγω ανεπαρκούς διασύνδεσης και το ίδιο ισχύει για το φυσικό αέριο. Μόνο 2% έχουμε στην περίπτωση αυτή και η ικανότητά μας για παροχή υγροποιημένου φυσικού αερίου θα μπορούσε να είχε βοηθήσει πάρα πολύ την Ευρώπη στην περίπτωση που ξεκινούσε μια κρίση στην παροχή φυσικού αερίου όπως είδαμε με την Ουκρανία πέρσι. Αλλά είναι απαραίτητο να αναπτύξουμε αυτές τις υποδομές αλλά όπως έλεγε και ο ο συναδελφό μου τα ισπανικά κόρτες υπάρχουν τόσο μεγάλες ε, διαφορές μεταξύ των χωρών μελών σε ό,τι αφορά το νομοθετικό πλαίσιο ώστε είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα την αποδεσμοποίηση και την διαφοροποίηση της διαχείρισης των δικτύων από τη μεταφορά ενέργειας από τα δίκτυα στην Ισπανία Έχουμε μια δημόσια επιχείρηση η οποία έχει φυσικό μονοπόλιο τόσο για την κατασκευή των υποδομών όσο και τη διαχείριση των ηλεκτρικών δικτύων. Νομίζουμε όμως ότι διατηρεί μια στάση η οποία είναι σωστή διότι επιτρέπει τη λειτουργία των δικτύων χωρίς να χρησιμοποιεί τη θέση της. Πιστεύω λοιπόν κύριε Κόβενη ότι θα ήταν απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι θα υπήρχαν οι διάφορες και συμμαχίες μεταξύ των εταιριών οι οποίες διαχειρίζονται τα συστήματα σε, ευρωπα... σε εθνικό επίπεδο ώστε να έχουμε δίκτυα που θα λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δίνω το λόγο στην συνάδελφό μου τώρα. Εγώ είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Βιομηχανίας ήδη. Ε, συμμετέχω για δεύτερη φοιτεία. Ως βουλευτής από τη Ρουμανία ίσως να έχω διαφορετικό πρίσμα και να βλέπω τα πράγματα από μια διαφορετική γωνιά. Όλα αυτά τα θέματα της ε, αγοράς ενέργειας. Καθώς δεν είμαστε ακόμη ε, μέρος της Ευρωζώνης. Η διασύνδεση ε, ιδιαίτερα ετέθη ως ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά τη μεγάλη κρίση για την προμήθεια σε φυσικό αέριο από την Ουκρανία προς την Βουλγαρία που ε, εξέθεσε στο ψύχος για ένα ολόκληρο χειμώνα κράτο μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είχε υποθεί λοιπόν τότε ότι αν υπήρχε κόμβο μεταξύ Βουλγαρίας και Ρουμανίας θα είχαμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τη Βουλγαρία να επαναπροσανατολίσει, να αλλάξει δηλαδή πορεία ενός, ε, ε, της παροχής του φυσικού αερίου από αλλού και να εξασφαλίσει, ε, εξασφαλιστεί ανάγκες της. Επίση υπήρξε μια πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με μια έκθεση του κυρίου Βιντάλ Κουάντρας για την ασφάλεια σε ε, προμήθεια ενέργεια. Η έκθεση του κυρίου Βιντάλ Κουάντρας ακόμη είναι κρεμής, είναι συζήτηση. Πάντως η ιδέα της διασύνδεσης των δικτύων προτείνεται ως υποχρεωτική και ίσως θα πρέπει να κρίνουν οι κυβερνήσεις να λάβουν τι αποφάσει του για τι επενδύσει. Δηλαδή θα πρέπει και τα κράτη-μέλη από, μέλη από πλευρά του να δεσμευτούν και να επιτελέσουν το καθήκον που του εμπίπτει ω προ την ε, ασφάλεια στην προμήθεια ενέργεια. Για δε τα κίνητρα για την οικονομία, δηλαδή για τις επιχειρήσεις, είναι ανοιχτό ζήτημα. Εγώ είμαι φιλελεύθερη, ανήκω στην ομάδα των φιλελευθέρων και ω εκ τούτου πιστεύω ότι χωρί κίνητρα η αγορά δεν μπορεί απαραίτητα να ανταποκριθεί σε αυτό που επιδιώκουν οι πολιτικοί. Θα ήταν ενδιαφέρον λοιπόν κάποιοι από εσά, με την εμπειρία που έχετε από τι χώρε σα να συμβάλλετε σε αυτέ τι ε, προτάσει και την ανταλλαγή απόψεων που διατυπώνονται ω προ την ε, παροχή κινήτρων για τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, ενδιαφέρον αυτό που είπατε εσείς για τις ε, κρατικές επιχειρήσεις και τις αντιδράσεις από ορισμένα τμήματα της αγοράς τους προς την διασύνδεση. Ακριβώς επειδή υπάρχει ζήτημα προστασίας της ε, θέσης τους μέσα στην εθνική αγορά. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα πρέπει να το λύσουμε το ζήτημα στο ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί μέσα σε κάθε κράτος μέλος χωριστά δεν μπορεί να λυθεί. Ένα βήμα θα ήταν αυτό. Να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη ε, να τηρήσουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια ως προς την προμήθεια, ως προς την ασφάλεια της προμήθειας ενέργειας. Δηλαδή διασύνδεση στο δίκτυο. Για δε τα βιοκαύσιμα, εγώ είμαι με, μεταξύ εκείνων που δεν πιστεύουν στην ε, ε, επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Πολλά είναι τα προβλήματα που διαπιστώνονται και μετά τον ε, το ενθουσιασμό που επικράτησε στην αρχή όταν εμφανίστηκε αυτή η εναλλακτική, βλέπουμε σε πολλές αγορές και ιδιαίτερα και στην Αμερικανική, στι ΗΠΑ δηλαδή, ότι φυσικά μπορείτε να έχετε και τις δικές σας αντιρρήσεις ασφαλώ, αλλά βλέπω εγώ τουλάχιστον ότι δεν βγάζει πουθενά αυτή η ιστορία με τα βιοκαύσιμα. Για την αποδέσμευση βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές ε, αντιδράσεις από ορισμένα κράτη-μέλη ως προς την πλήρη αποδέσμευση. Και γι' αυτό βλέπουμε κάποια μείγματα, δηλαδή διαχείριση του unbundling και όχι, μάλλον ε, unbundling αποδέσμευση όπως τη διαχείριση και όχι ως προς την ιδιοκτησία. περιπτώσει, αυτό νομίζω όμως ότι δεν χρειάζεται να μας οδηγήσει σε μια νέα συνθήκη. Όσο ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί οι ισχύοντες κανόνες. Αυτό είπα και στην αρχή της ομιλίας μου. Υπάρχει νομοθεσία και όμως δεν εφαρμόζεται. Ας εφαρμοστεί λοιπόν πρώτα αυτή η νομοθεσία. Και για τον εκπρόσωπο της ECB θα ήθελα να ρωτήσω και ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση που μας κάνατε. Αλλά ήθελα να ρωτήσω το εξή. Όλο αυτό το ζήτημα μπορείτε να το ενσωματώσετε στην προοπτική της παγκόσμιας αγοράς, δηλαδή η θέση της ευρωπαϊκής αγοράς μέσα στην παγκόσμια και αντίκτυπος του δολαρίου στην δική μας ενεργειακή αγορά. Ξέρουμε ότι γενικά οι συναλλαγές στην ενέργεια αναπτύσσονται σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε εμεί το νόμισμα στο οποίο γίνονται οι συναλλαγέ. Και γι' αυτό το λόγο και θα ήθελα να μα πείτε πώ βλέπετε στα πράγματα και πόσο επηρεάζει το δολάριο την εσωτερική μα αγορά στην ενέργεια. Κύριε Ρόφερ. Ευχαριστώ, πολύ. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια ως προς τα στοιχεία που έχουμε και από την έκθεση. Καταρχάς ως προς την διασύνδεση. Βλέπουμε στην έκθεση ότι όντως, χωρίς να είναι βέβαια η κατάσταση, η ασφάλεια στην ενέργεια, χάρη στην διασύνδεση των αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με τη δεκαετία του 90, Φερρυπίν. Δεν μπορούμε να λέμε δηλαδή ότι δεν έχει γίνει τίποτα στον τομέα αυτόν. Και βέβαια ε, έχουμε πλεονέκτημα συγκρινόμενοι με τις ΗΠΑ στο θέμα της διασύνδεσης. Αλλά φυσικά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και θα συμφωνήσετε και εσείς πιστεύω ότι πρόκειται πάνω απ' όλα για στοιχείο της ασφάλειας των προμηθειών μας ενέργεια. Γι' αυτό πάνω απ' όλα πρέπει να ενισχύσουμε την διασύνδεση. Για δε την αποδέσμευση, το unbundling, υπάρχει αφενός, υπάρχουν διάφορες πτυχές. Υπάρχει αφενός το περιθώριο κέρδους που μπορούμε να υπολογίσουμε εφόσον ε, έχουμε αυτή την ενοποίηση της αγοράς. Αφετέρου όμως υπάρχουν κάποιοι οποίοι πιστεύουν ότι η ενοποίηση και στην παραγωγή και στη διανομή μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα της διαδικασίας παραγωγής και διανομής συνολικά. Έτσι και στην πορεία της απελευθέρωσης των αγορών διαπιστώνουμε ότι η αποδέσμευση ή η φιλελευθερωποίηση βοηθάει να πέσουν οι τιμές. Άρα έχει νόημα να κάνουμε προσπάθειες περισσότερο για το στοχό αυτόν. Έχουμε δηλαδή απτά στοιχεία που μας πείθουν ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Για τα βιοκαύσιμα, εμείς δεν έχουμε να δώσουμε συγκεκριμένη απάντηση. Αν δείτε τα πιθανά σενάρια που προτείνονται ως προς τις μελλοντικέ εξελίξεις για τον χώρο του ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Διεθνή Οργάνωση Ενέργειας, βλέπουμε περισσότερη ε, πιο έντονη συμμετοχή στο μείγμα των ανανεώσιμων πηγών, αλλά πάντως πάλι περιορισμένη συμμετοχή, περιορισμένα ποσοστά και ε, διατήρηση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Η τελευταία σας ερώτηση για το συσχετισμό δολαρίων ΗΠΑ και ενεργειακών τιμών. Ναι, όντως, διαπιστώνεται ότι υπάρχει ευθεία συνάρτηση μεταξύ των ισοτιμιών και των τιμών της ενέργειας, η οποία όμως δεν είναι πάντοτε σταθερή. Άρα δεν είναι δεδομένο ότι το αποτέλεσμα είναι πάντα στην μία κατεύθυνση. Και ως εκ τούτου δεν είναι δεδομένη η σχέση της διακύμανσης του δολαρίου με τις διακυμάνσεις τιμές ενέργειας. Και γι' αυτό και δεν είναι δεδομένοι οι όροι υπό τους οποίους μπορούν να εγγραφούν ως οικονομικές ε, μονάδες οι τιμές ενέργεια στις παγκόσμιες αγορές. Το είδαμε εν μέρη να, να υπάρχει, είδαμε ότι υπήρχε μια ευθεία συνάρτηση με το δολάριο στη τελευταία μεγάλη ενεργειακή κρίση, αλλά δεν είναι πάντοτε δεδομένο ότι η ισοτιμία θα ε, οδηγήσει σε αύξηση των ενεργειακών τιμών. Επίσης, οι σημαντικές διακυμάνσεις στις μέσες ενέργειας που είδαμε το 2008-2009 οφειλόταν και σε διαφορετικές συνθήκες προσφοράς και ζήτησης. Δεν μπορούμε λοιπόν την ισοτιμία να την κατηγορήσουμε ως αποκλειστική υπέτειο των διακυμάνσεων στις τιμές ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Τα τέσσερα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν <clears throat> αναφέρονται πρώτα απ' όλα στα δίκτυα. Η διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων έχουμε είδαμε ότι στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών αυτός ο οποίος έχει το, την κατοχή του δικτύου μπορεί θαυμάσια να εξασφαλίσει τη λειτουργία του δικτύου και να υπολογίσει το τίμημα το οποίο θα πρέπει να καταβάλει ο χρήστης αυτού του δικτύου. το ίδιο μπορεί να γίνει και στην περίπτωση της ενέργειας έχουμε μιλήσει, δεύτερο ερώτημα, μιλήσαμε για τις βιώσιμες, τις ανανεώσιμες ενέργειες. Τι σημασία μπορεί να έχει λοιπόν κάθε ενέργεια, αυτό οφείλεται και στους όρους παραγωγής της κάθε ενέργειας και στην τεχνολογία που υποστηρίζει αυτή την παραγωγή. Μέσα στην Ευρώπη λοιπόν υπάρχει δυνατότητα και ενοτομία και τεχνολογική εξέλιξη. Μπορούν να υπάρξουν χώρε οι οποίε θα θέλουν να ε, ειδικευτούν σε, στην παραγωγή ορισμένων ειδών ενέργεια. Ορισμένε χώρε στην αιωλική ενέργεια, άλλες να αφορούν ε, βιώσιμο, βιοκαύσιμο παραγωγός χάρη κάτι άλλο και τελικά να, τα τελικά αποτελέσματα να αντανακλούν την ισορροπία μεταξύ αυτών των ειδών ενέργειας. Για το θέμα της, των επιχειρήσεων νομίζω το απήντησα με το πρώτο ερώτημα. Τέταρτο, για να μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα στο τωρινό πλαίσιο, πρέπει πράγματι να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το πλαίσιο, να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα και όχι να δημιουργήσουμε περαιτέρω προβλήματα τα οποία μας, επι... υποχρεώνουν να αναζητήσουμε νέες λύσεις. Εγώ δεν νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου οι πολίτες έχουν την δυνατότητα ελεύθερης διακίνησης, όπου υπάρχει μια κοινή αγορά αγαθών, η ενέργεια που κανονικά δεν έχει σύνορα να πρέπει να περιορίζεται μέσα στα εθνικά σύνορα. Γιατί αυτό περιορίζει πάρα πολύ την ε, ανάπτυξη των ανανεωσίμων ενεργειών. Γιατί αν μια χώρα μπορεί να παράγει ανανεώσιμε ενέργειε, παραδείγματο χάρη αιωλική ενέργεια καλύτερα από τι άλλε χώρε, μπορεί αυτή η ενέργεια να χρησιμοποιηθεί από άλλε χώρε. Οι τεχνολογικέ λοιπόν πρόοδοι που γίνονται σε μια χώρα για μια συγκεκριμένη μορφή ενέργεια μπορούν να βοηθήσουν όλε τι χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εκμεταλλευτούν αυτή την πρόοδο. Γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει και παγκόσμιο επίπεδο είναι απαραίτητο σε παγκόσμιο επίπεδο να υπάρξει βιώσιμη παραγωγή ενέργεια γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για τη διατήρηση τη ζωή στον πλανήτη μα. Γι' αυτό η Ευρώπη θα πρέπει να δώσει τι απαντήσει σε αυτή την αδύρυτη ανάγκη να βρούμε λύσει για την ενέργεια. Κυρία κυρία Νιουθορκίσα, σα ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Κόβενη. Έφυγε δυστυχώ ο κύριο Κόβενη που μας είχε λείψει τόσο μετά που έφυγε από την προηγούμενη θητεία αναφερόμαστε στα τροτά σημεία της Ευρώπης και το γεγονός ότι είναι εύθραστη η Ευρώπη και εξαρτάται από ορισμένου ε, παρόχους ενέργειας που είναι ασταθείς όπως είναι οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, Ρωσία, Ουκρανία κτλ. Και κινδυνεύουμε να συνάψουμε συμφωνίες με χώρες στις οποίες είναι ακόμα λιγότερο αξιόπιστες όπως είναι το Τουρκμενιστάν και άλλες. Είναι απαραίτητο λοιπόν να έχουμε σχέδια τα οποία θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια τροφοδοσίας όπως είναι το σχέδιο Ναμπούκο για να μπορούμε να έχουμε σταθερή παροχή φυσικού αερίου και πετρελαίου. Επίσης, παράλληλα με την ανασφάλεια που υπάρχει στις πηγές, ποτέ δεν μιλάμε για την πραγματική αυτόχθονο πηγή, αυτόχθονα πηγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ο άνθρακος που έχει δαιμονιοποιηθεί λόγω της ανάγκης να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος αλλά που με τις ε, νέες τεχνολογίες όπως είναι η συγκράτηση και αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακος μπορεί πράγματι ο άνθρακας να λειτουργήσει και να είναι πηγή νέων τεχνολογιών και παραγωγής ενέργειας. <clears throat> Επομένως πιστεύω κάπου πρέπει να αναφέρεται και στα έγγραφά μας το θέμα της χρησιμοποίησης του ενδογενούς άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον αυτή η πηγή που βρίσκεται στην Ευρώπη ο άνθρακας θα ληφθεί υπόψη όταν εμείς σχεδιάζουμε για την ενεργειακή Ευρώπη στο μέλλον. Όπως είπε και ο κ. Λαβίγια, είναι πάρα πολύ σημαντική η διασύνδεση και είναι απαραίτητο να έχουμε <clears throat> μια, ε, ένα διαμοιρασμό των ανανεώσιμων ενεργειών και να έχουμε μια κοινή αγορά για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, ίσως θα πρέπει να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις και να υπάρχουν ομοδοποιημένες απαντήσεις. Ο κύριος Βόρης ζήτησε το λόγο επίσης από την Λιθουανία. Κυρία Ράουκο μετά. Α, εδώ είναι, εδώ είναι, συγγνώμη. Έχω την αίσθηση ότι και στη δική μου χώρα, όπως και στην περίπτωση της Ιρλανδίας, αυτό το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο είναι οι διασυνδέσεις. Έχουμε μια εξαιρετική, βιώνουμε μια εξαιρετική σε εισαγωγικά κατάσταση. Είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι από μια ουσιαστική πηγή, δηλαδή τη Ρωσία και αυτό αφορά και τον άνθρακα και το φυσικό αέριο. Δεν έχουμε ουσιαστικά καμία σύνδεση με τα δίκτυα διανομής ενέργειας της Δυτικής Ευρώπης. Το 2009 το σχέδιο διασύνδεσης το οποίο έγινε δεκτό από το Λιθουανικό Κοινοβούλιο θα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις απομόνωσή μας της ενεργειακής, να αποκαταστήσουμε δικτυώσεις με τις γειτονικές χώρες. Ελπίζω τα σχέδια τα ευρωπαϊκά να αστραφούν και αυτά προς την κατεύθυνση την ίδια από την οποία εμείς ακολουθούμε και να μπορέσουμε να συνδεθούμε και με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Μόνο μέσα από αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση μέσα στην οποία κινούμεθα και θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε λογικές τιμές για τους ε, καταναλωτές μας. Δεν ξέρω αν μπορούν να με βοηθήσουν εδώ οι εμπειρογνώμονες, δεν ξέρω αν χωρίς την ενιαία αγορά σαν παράδειγμα μπορούμε να φτάσουμε στους στόχους τους οποίους θέλουμε. Κύριε Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω την παρέμβασή μου Υπενθυμίζω, υπενθυμίζουσα καλύτερα, αυτό το οποίο ήταν το πολύ καλό παράδειγμα της Πορτογαλίας και της ε, Ισπανίας για τη δημιουργία μιας κοινή αγοράς ιβυρικής ενέργειας. Επίσης, σε ό,τι αφορά την αποδεσμοποίηση, η Πορτογαλία και η Ισπανία έπαιξαν πρωτοπόρο ρόλο στη δημιουργία μιας απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας και επομένως η Ευρώπη ακολούθησε το δικό μας παράδειγμα και όπως είπε και ο Ιρλανδός συναδελφός μας προσπαθεί ακόμα να ακολουθήσει το βέλτιστο παράδειγμα που έδωσε η Ισπανία και η Πορτογαλία. Επίσης η Πορτογαλία ακολουθώντας μια πολιτική αηφόρο ενέργεια Έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες, έχει αναγνωριστεί το γεγονός ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη επένδυση σε αιωλική και ηλιακή ενέργεια, ιδίως στην Πορτογαλία. Είμαστε σε μεγάλο βαθμό ηγέτες σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ό,τι αφορά κυρίως την αιωλική ενέργεια και ένα δίκτυο ανανεώσιμων ενεργειών στην ε, Ευρώπη θα βοηθούσε ιδιαίτερα την Πορτογαλία, η οποία εξάγει ήδη τεχνολογία προς άλλες χώρες, παράγει ε, υλικά και εξοπλισμό αιωλικής ενέργειας και είναι σε θέση να εξαγάγει αυτά τα προϊόντα, επομένως ένα δίκτυο για την αιωλική ενέργεια, γενικά για, την, ε, για τις ανανεώσιμες ενέργειες θα ήταν πολύ θετικό. Επίσης πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δημόσιες, ε, τους δημόσιες προμήθειες, τους δημόσιους διαγωνισμούς σε ό,τι αφορά την ε, ενέργεια όταν ανανεώνουμε παραδείγματος οι υποδομές. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω και κάτι σε σχέση με τις δομές, με τη διάρθρωση μάλλον της τιμολόγηση της ενέργειας. Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι οι εταιρείε πετρελοειδών που όταν αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου, του αργού πετρελαίου, παρακολουθούν πολύ γρήγορα την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, ενώ όταν κατεβαίνουν οι τιμές Εκεί είναι πραγματικά βραδία η προσαρμογή τους και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να το εξηγήσει κανείς, πολύ λιγότερο να το αποδεχθεί ότι ο πολίτης τελικά πληρώνει πιο ακριβά το βαρέλι του πετρελαίου. Εμεί πιστεύουμε ότι το γεγονός ότι οι τελικές τιμές του καταναλωτή ενώ δεν καλύπτονται από συγκεκριμένα εργαλεία για να τις ε, προστατεύει κανείς είναι πολλές φορές αντικείμενο κοινών προσπαθειών των εταιριών για να μείνουν σε υψηλό επίπεδο και προσπαθούν να κερδίσουν πάντα όλο και περισσότερα <clears throat> από την τιμή στον τελικό καταναλωτή. Θέλω λοιπόν να καταθέσω αυτή τη μαρτυρία ότι για μας η δημοκρατικοποίηση της πρόσβασης στην ενέργεια και το δίκαιο τίμημα της ενέργειας θα πρέπει να είναι όχι μονάχα μια αναγκαιότητα αλλά και μια πραγματικότητα. Η χώρα μας ήταν ψηφιακή, πέρασε στο ψηφιακό επίπεδο με το πρόγραμμα Μαγκελάνος πολύ πιο πριν από άλλες χώρες της Ευρώπης. Από την ε, πρώτη τάξη του Δημοτικού δηλαδή ήδη έχουν τον υπολογιστή τους, έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Επομένως η Πορτογαλία έχει ευνοηθεί πάρα πολύ από τη δημοκρατικοποίηση της πρόσβασης στα δίκτυα πληροφορικής και το ίδιο θα γίνει και στην περίπτωση ενέργειας. Είναι απαραίτητο λοιπόν για την ηλεκτρική ενέργεια και το λέω αυτό γιατί μία, ένα από τα παράπονα που ακούμε πολλές φορές από τους Πορτογάλους βιομηχάνους είναι ότι η βιομηχανία μας δεν καταφέρει να είναι πιο ανταγωνιστική από την Ισπανική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ισπανική κυβέρνηση επιδοτεί το κόστος του βιομηχανικού ηλεκτρισμού και επομένως υπάρχει ένα τεχνητά χαμηλό κόστος. Αυτό όταν γίνεται μονάχα σε μια χώρα φανταστείτε πόσο πιο δύσκολο θα είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν υπάρχουν επιδοτήσεις. Από την άποψη αυτή λοιπόν σας λέω και πάλι ότι η ενέργεια είναι ένα εγκάρσιο θέμα, ένα θέμα που έχει κοινωνικές πτυχές, έχει να κάνει με την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα κάθε χώρας και θα ήθελα να επικεντρώσω την δική μου προσοχή στο θέμα αυτό των εργαλείων που μπορούν να βοηθήσουν την Ευρώπη να παίξει πρωτοπόρο ρόλο στα θέματα αυτά χωρίς να θίξουμε βέβαια τη δική μας ανταγωνιστικότητα και αυτά ήθελα να πω προς το παρόν. Ωραία, μπορούμε να κλείσουμε με τον κύριο Εσκέδα από την Ισπανική Γερουσία. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Φελισλαρία και τον κύριο Ρόλ για την ε, μελέτη που παρουσίασε που είναι πολύ ενδιαφέρουσα από πολλές πτυχές. Θα ήθελα επίσης να βγει και κάποιο συμπέρασμα από όλα αυτά τα πράγματα που είπατε, γιατί υπάρχει απόκληση των τιμών, όχι μόνο της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά γενικά των πηγών ενέργειας όταν υπάρχουν παρόμοιες πηγές με παρόμοια διάρθρωση κόστους. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τύχουν κάποιες εξήγησεις. Τώρα, οι τιμές της ενέργειας γενικά, αν μπορούσαμε να έχουμε διασύνδεση των δικτύων ενέργειας σε όλη την Ευρώπη, θα είχαμε ένα είδο συγκοινωνούντων δοχείων και θα μπορούσαν να εξισω... εξισωθούν σημαντικά οι τιμές. Αλλά τώρα όταν έχουμε επιχειρήσεις ιδιαίτερα ισχυρές οι οποίες δραστηριοποιούνται στις χώρες μας και πολλές φορές η ίδια χώρα δραστηριοποιείται σε πάρα πολλές χώρες αντιμετωπίζουμε πολλά θέματα τα οποία ανακύπτουν. Όλες οι επιχειρήσεις είναι ίσες, αλλά κάποιες είναι λιγότερο ίσες από τις άλλες. Υπάρχει πάντως ένα παράδειγμα στην Ευρώπη, κάτι το ενός ε, πολύπλοκου θέματος το οποίο έχει επιληθεί. Είναι ένα από ένα άλλο τομέα βέβαια αυτό. Είναι τα θέματα των τρένων. Όλες οι χώρες έχουν διαφορετική νομοθεσία Όλες οι χώρες έχουν διαφορετικά έθιμα, όλες έχουν πολλές φορές και διαφορετικό εύρος γραμμών και παρόλα αυτά αυτή τη στιγμή συγκεντρώνουν τις προσπάθειές τους για να υπάρχει μια καλύτερη διασύνδεση τρένων από τη μία άκρη της Ευρώπης ως την άλλη. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η προσπάθεια αυτή, είναι ένα τεράστιο σχέδιο στο οποίο γίνονται τεράστιες προσπάθειες για τη διασύνδεση του βορείου τμήματος της Ευρώπης με τον νότιο, ανατολικού και δυτικού και επίσης υπάρχει το θέμα αυτό το οποίο έχει καθυστερήσει πάρα πολύ να υπάρξει δυνατότητα παραγωγής ηλιακής ενέργειας στη Σαχάρα και να έρχεται στη Βόρεια Ευρώπη μετά από εκεί. Αλλά υπάρχει μια ομοιότητα μεταξύ αυτών των σχεδίων και όλους αυτούς τους λόγους νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ όλων των χωρών για να προωθηθούν αυτά τα σχέδια. Τώρα, η επέκταση της διασύνδεσης θα μπορούσε να εξισώσει την τιμή της ενέργειας. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι έχουμε να κάνουμε με εταιρείε οι οποίες είναι ιδιαίτερα ισχυρές και με τον τρόπο αυτό τροχοπεδούν την προσπάθεια να υπάρξει νομοθεσία η οποία θα ευνοήσει με τον καταναλωτή αλλά όχι αυτές τις εταιρείε. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη ρύθμιση των αγορών με νομοθετικά μέτρα και από όλα αυτά τα στοιχεία το πιο επικίνδυνο για μένα είναι να μην λάβει κανείς τους καταναλωτές γιατί κανείς δεν έχει μιλήσει εκτενώς για τους καταναλωτές. Θα πρέπει να οικοδομήσουμε την Ευρώπη, θα πρέπει η Ευρώπη τουλάχιστον να εξασφαλίσει ότι έχουμε ασφάλεια κατανάλωσης. Να μην ξαναγίνει αυτό που είχε γίνει στην κεντροανατολική Ευρώπη με το φυσικό αέριο. Να είναι επίσης προσβάσιμο το τίμημα της ενέργειας για τον καταναλωτή και η ενέργεια αυτή να είναι όσο το δυνατόν πιο καθαρή. Δεν θα πω τώρα στι λεπτομέρειε πώ θα γίνει αυτό, αλλά θα πρέπει να κινηθούμε προ την πιο καθαρή δυνατή μορφή ενέργεια, γιατί θα πρέπει να διασώσουμε και τον κόσμο. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο έλεγχο των εταιριών και να μην έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν υπερβολικά δεσπόζουσε θέσει και να σέβονται και τον ανταγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ. Bueno, hay muchas, eh, Υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί. Η κυρία Βαλεάν ίσως μπορεί να αρχίσει να απαντά, να δώσει μια πρώτη απάντηση. Πολύ ευχαριστώ να σχολιάσω στις παρατηρήσεις που ακούστηκαν. Αν και δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι είμαι ειδική. Πολιτικός είμαι μόνο, όπως και εσείς και προσπαθώ να καταλάβω ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές που μας υποδεικνύουν οι πραγματογνώμονε. Νομίζω ότι υπάρχει ήδη ένα συμπέρασμα, το ζήτημα της διασύνδεσης καταρχάς. Το επισημαίνουν οι πάντε ως άκρος απαραίτητο, ως απολύτως απαραίτητο για την βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας. Διασύνδεση λοιπόν, διασυνδέσεις. Όπως όμως εσείς επισημάνατε, Υπάρχουν και τα εθνικά συμφέροντα, τα οποία αντιτίθενται στην ανάπτυξη, στην οικοδόμηση αυτής της ενιαίας αγοράς εργασίας. Εθνικά συμφέροντα τα οποία ε, υποστηρίζουν τις εθνικές επιχειρήσεις. Όντως, και όπως είπατε και εσείς πολύ εύστοχα, δεν είναι πρώτο μέλημα αυτών των συμφερόντων το συμφέρον του καταναλωτού. Συμφωνώ απολύτως ότι θα έπρεπε να υπάρχουν απελευθερωμένες αγορές. Χωρίς απελευθερωμένες αγορές δεν νοείται μείωση των τιμών και επικοινία στην προμήθεια, στο μείγμα προμήθειας. Δεν ξέρω πώς μπορεί να επιληθεί το ζήτημα αυτό, γιατί είναι πολλές οι χώρες οι οποίες προσφέρουν επιδοτήσεις. Η δική μου η πατρίδα, παραδείγματι, και από την άλλη πλευρά ξέρω ότι και οι Βρυξέλλες προσπαθούν να πιέσουν για την απελευθέρωση των αγορών. Ε, αλλά με δεδομένη την μεγάλη οικονομική κρίση και τα, τα πλήγματα που έχουν υποστεί οι καταναλωτές ε, είναι ίσως δύσκολο να καταργηθούν στην τωρινή στιγμή οι επιδοτήσεις αυτές. Για το ζήτημα του Ναμπούκο μείωση της εξάρτησης από τη μία πηγή Ε, δεν εξασφαλίζεται όταν προσπαθούμε να κατασκευάσουμε αγωγούς που περνούν πάντα από την ίδια πηγή. Είμαι επιφυλακτική απέναντι στον Αμπούκοκο Γιατί δεν ε, έχω καμιά ένδειξη ότι κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα θα γίνει ξαφνικά. Θα αρχίσει τώρα εάν πραγματοποιηθεί το Ναμπούκο όπως έχει σχεδιαστεί μέχρι τώρα. Τώρα αν κάτσει κάποιος κάτω και, σοβαρά, με σοβαρότητα ε, ξαναχαράξει την πορεία του φυσικού αερίου, τον αγωγό δηλαδή, τότε ναι μπορεί Ίσως το παράδειγμα της ε, Ισπανίας να είναι χρήσιμο γιατί η Ισπανία είναι τόσο μακριά από τη Ρωσία που δεν ε, μπορεί να στηριχθεί στη λειτουργία αγωγών. Έχει λοιπόν κατασκευάσει θερματικούς σταθμούς φυσικού αερίου στους οποίους καταφθάνει φυσικό αέριο από ολόκληρο τον κόσμο και όχι μόνο από μία πηγή. Αν λοιπόν έχουμε ένα δίκτυο ε, θα μπορούσαμε με ένα και μόνο σημείο εισόδου να διανέμουμε το αέριο σε διάφορες κατευθύνσεις. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι θα το καταφέρουμε αυτό. Αυτά προς το παρόν. Και εγώ θα ήθελα καταρχήν να απαντήσω την κυρία Μουνή Θορκίσα. Είπα στην αρχή όταν ε, λάβα το λόγο για πρώτη φορά ότι η τεχνολογία θα προκαθορίσει σε μεγάλο βαθμό την ε, πορεία κάθε ενεργειακής πηγής. Ο άνθρακας είναι μια αυτόχθον πηγή στην Ευρώπη, θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε αυτή την πηγή και υπάρχουν πράγματι τα προγράμματα αυτά συγκράτησης και αποθηκεύσης διοξιδίου του άνθρακος και υπάρχουν και προγράμματα για την καθαρή εκμετάλλευση του άνθρακος ή την τεχνολογία καθαρής καύσης. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, όχι μόνο για μία πηγή αλλά για όλες τις πηγές και μια ευρωπαϊκή χώρα από μόνη της είναι πολύ δύσκολο να έχει αρκετά χρήματα για να αναπτύξει τις ε, ανανεώσιμες ενέργειες και τις καθαρές ενέργειες. Αλλά όλες οι χώρες από κοινού είναι υποχρεωμένες να το κάνουν. Εγώ τονίζω ιδιαίτερα αυτό το τομείο γιατί δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο. Δεν πρόκειται για την... Ε, ε, ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης αλλά για την πρωτοπορία της στην δημιουργία απασχόλησης και στην τρίτη αυτή βιομηχανική επανάσταση που θα λάβει η χώρα στον κόσμο στα ενεργειακά θέματα. Αν χάσουμε την πρωτοπορία και την ηγεσία σε ό,τι αφορά τεχνολογική έρευνα για τα θέματα ενέργειας, τότε όχι μονάχα θα έχουμε προβλήματα με την ενεργειακή τροφοδοσία των Ευρωπαίων, αλλά θα γίνουμε πια ουραγοί σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά τα θέματα της ενέργειας, κάτι το οποίο θα μας στήξει τα μάλα σε αυτή την τεχνολογική επανάσταση και η επανάσταση αυτή η τεχνολογική μπορεί να είναι εξόδου από την οικονομική κρίση την οποία διατρέχουμε και το υβηρικό, η υβηρική αγορά η κοινή αγορά ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν έχει λοιπόν σύνορα η ενέργεια θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί να κινείται ελευθέρως σε ένα συμπεφωνημένο πλαίσιο. Έχουμε επιλύσει πολύ πιο δύσκολα προβλήματα. Υπάρχουν δυσκολίε, αλλά μπορούμε να τις υπερπηδήσουμε. Γιατί χωρίς καμία αμφιβολία ακόμα και μια χώρα η οποία θα θεωρήσει ότι θίγεται από την κοινή λύση πάλι θα έχει τεράστια πλεονεκτήματα. Θυμάμαι στην περίπτωση της Καστήλης στην ε, Ισπανία πριν από την ε, ανακατανομή, πριν από τον αναδασμό, την ανακατανομή των αγροτεμαχίων ήταν ιδιαίτερα κατακαιρματισμένη η κλήρη. Λοιπόν, με, την, με τον αναδασμό μπόρεσε να απογειωθεί η γεωργία και να προχωρήσει πολύ γρήγορα. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι θεωρούσαν ότι έχαναν από την άποψη αυτή, γιατί είχαν τα καλύτερα αγροτεμάχια, καταφέραν να αποκομίσουν τα ε, πλεονεκτήματα τη συνεκτικότητα των ε, αγροτεμαχίων τους. Αυτό οδήγησε σε μεγαλύτερη παραγωγή, καλύτερη ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Λοιπόν, σε τελική ανάλυση οδήγησε σε ωφέλη για όλους. Για αυτά που είπε ο κ. Σισκέδα για την απόκληση των τιμών και της και τις διασυνδέσεις, ναι. Αν έχουμε μια ενιαία αγορά μπορούν να είναι πιο ενιοποιημένες οι προδιαγραφές, να έχουμε κοινού κανόνες του παιχνιδιού και αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Το είδαμε αυτό στα τρέλα και μπορούμε να το δούμε και στις, ε, στους τομέα της ενέργειας. Ο καταναλωτής λοιπόν θα έχει τη δυνατότητα να έχει την ε, πρόσβαση στην ενέργεια από όπου και να προέρχεται και αυτό είναι απαραίτητο για τον 21ο αιώνα. Θα βοηθήσει τους, Ευρώπου, ε, τους πολίτες να καταλάβουν ότι η Ευρώπη είναι ισχυρή και μπορεί να δίνει λύσεις στους πολίτες. Μάλιστα. Πάρα πολύ σύντομα η ανησυχία στην οποία αναφερθήκατε για τους καταναλωτές. Προσπάθησα να το πω και εγώ στην εισαγωγή μου. Το βασικό μας θέμα είναι αυτό. Γι' αυτό εξετάζουμε την τιμή στον καταναλωτή κυρίως και πριν από κάτι άλλο. Υποστηρίζω λοιπόν την προοπτική αυτή. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο σημαντικές για τα σχόλια. Για το θέμα της ασημετρίας. Γνωρίζετε ίσως καλύτερα από μένα φυσικά, σίγουρα καλύτερα από μένα το τι συμβαίνει στην Πορτογαλία. Ποια είναι τα μέτρα που λύθηκαν... και ποιες οι αντιδράσεις. Αλλά τουλάχιστον για τις εξελίξεις τη τιμές από πάνω προς τα κάτω, εμείς δεν βρίσκουμε κάποια στοιχεία στις διάφορες χώρες και στη δική σας χώρα. Ίσως να υπάρχει μια κάποια χρονική υστέρηση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν διαπιστώσαμε μια συστηματική ασυμμετρική τάση όταν υπάρχει μείωση των τιμών ενέργειας. Μπορεί να υπάρχουν κάποια μικρά λάθη στην αξιολόγηση αυτή, αλλά οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην κρίση μας σχετικά με τις επιδοτήσεις. Θα συμφωνήσω ότι όταν οι επιδοτήσεις αυτές οδηγούν σε στρεβλώσεις της αγοράς αυτό είναι σαφέστατα αντιπαραγωγικό. Το θέμα είναι να προσπαθήσει κανείς να δημιουργήσει μακροπρόθεσμες προοπτικές και αυτό γιατί η ενέργεια και τα δίκτυα της ενέργειας απαιτούν βαρύτατες επενδύσεις και από αυτή την άποψη θα πρέπει να ακολουθούνται συνεκτικές πολιτικές και με διάρκεια σε επίπεδο λήψης πολιτικών αποφάσεων και στα πλαίσια προβλημάτων όπως η αντιμετώπιση του ε, αερίου των θερμοκηπίου. και σε σχέση με τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την βοήθεια στην κάλυψη του κόστους της ενέργειας ή στην επιδότηση ορισμένων τμήματων αυτής σχετικά με την απελευθέρωση των αγορών για το αν θα έπρεπε να υπάρχουν παντού ίδιες τιμές στα διάφορα επίπεδα είτε στην πηγή αυτό είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί στις Ηνωμένε Πολιτείες σαν παράδειγμα βλέπουμε ότι το μίξ της ενέργειας το οποίο χρησιμοποιείται αναχώρα για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος είναι εντελώς διαφορετικό. Σε μια χώρα το ποσοστό της πυρηνικής ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρισμού είναι ιδιαίτερα υψηλό, σε άλλες χώρες είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Οπότε η αύξηση της τιμής του πετρελαίου επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο την αύξηση της τιμής του προϊόντος σε κάθε χώρα. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους διαφέρουν οι τιμές. Το άλλο θέμα είναι το δίκτυο, το κόστος των δικτύων. Το κόστος των δικτύων είναι εντελώς διαφορετικό από χώρα σε χώρα. Υπάρχει το θέμα του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός όσο πιο αυξημένος είναι τόσο χαμηλότερες είναι οι τιμές. Αν θέλει κανείς να λάβει το λόγο, εάν θέλει, θέλω να πω τρία πράγματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να τα τονίσουμε. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι έχουμε τονίσει τη σημασία της, πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της ενεργειακής εξοικονόμησης, να υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη αποδοτικότητα και μεγαλύτερη εξοικονόμηση της ενέργειας. Δεύτερον, θα πρέπει να, θεωρηθού, να θεωρηθεί η ενέργεια σημαντική εισρωή όχι μόνο για τους καταναλωτές αλλά και για την βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα της υπήρου μας, όχι μονάχα στην μεταποίηση, όπου είναι σημαντική ενέργεια, αλλά όπως είπαν και οι συναδελφοί μου, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια τρίτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία βασίζεται και στην εξοικονόμηση και τις ε, καθαρές ενέργειες, όπου η Ευρώπη πρέπει να είναι πρωτοπόρος. Για τις διασυνδέσεις επίσης η Ισπανία έδειξε ότι αν είχαμε καλές διασυνδέσεις θα μπορούσαμε να δώσουμε και στην ε, Γαλλία και από εκεί στις άλλες χώρες της Ευρώπης φυσικό αέριο, θα μπορούσαμε να έχουμε μια πολύ καλύτερη συνεργασία για να αποτρέψουμε το κύμα ψύχους που πέρασε η Κεντρική Ευρώπη λόγω του, της διακοπής τροφοδοσίας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Λαβίγια. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους σας για τις ε, για τη συμβολή σας σε τόσο σημαντική αυτή η συζήτηση. Θα προσπαθήσουμε να τις συνοψίσουμε για το έγγραφο το οποίο θα παρουσιάσουμε αύριο στην Ολομέλεια. Όλα αυτά και ευχαριστώ πολύ. Τα είπανε, τα είπανε, τελειώσανε.